Σας καλωσορίζω και να καλωσορίσω και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράκη λόγω χρονικών περιορισμών. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία εισήγηση και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Θα πρέπει επίσης να συντομεύσουμε ελαφρώς το δεύτερο τμήμα που είναι οι ερωταπαντήσεις και να ομαδοποιήσουμε το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Πρόεδρε Ντράγκη, λοιπόν, ορίσατε Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο για την πρώτη ακρόαση φέτος ενώπιον της Επιτροπής σας. Τα δύο θέματα που επιλέξατε για τη σημερινή συζήτηση είναι εξαιρετικά επίκαιρα και αυτά θα συζητήσουμε. Καταρχάς, τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και δεύτερον τη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και τιμών καθώς και την τιμή αναφοράς για την νομισματική πολιτική. Ε, κάνοντας αυτό θα εξηγήσω γιατί η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσει δυνητικούς κινδύνους σε ένα περιορισμό μένο αριθμό τομέων που είναι κρίσιμη από την προοπτική ε, της ε, εντολής της για την πολιτική που πρέπει να ασκήσει. Άρα λοιπόν πρώτα ε, η, ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Είπα νωρίτερα στην ορμέλειά φέτος ότι η ευρωπαϊκή οικονομία ε, μεγεθύνεται στεναρά. Η μεγέθυνση είναι πιο σημαντική από ό,τι αναμενόταν σε διάφορους τομείς, σε όλους τους τομείς ε, σε μεγαλύτερο ρυθμό από ότι τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση. 2,5% μεγέθυνση είχαμε το 2017 στην Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλη εγχώρια κατανάλωση και επενδύσεις. Αυτές οι θετικές εξελίξεις έχουν προωθηθεί και στηριχθεί μέσω της, ε, των μέτρων ε, νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σημαντικά διευκόλυναν, χαλάρωσαν ε, τις συνθήκες δανεισμού για τα ενοικοκυριά και για τις εταιρείε, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν από τα μέσα του 2014 και του Οκτωβρίου του 2017, ο συνολικό αντίκτυπο στην μεγέθυνση τη Ευρωζώνης και του πληθωρισμού εκτιμάται και στι δύο περιπτώσεις να είναι 1,9% ορευτικά για την περίοδο 2016 με 2020 τα μέτρα μας ε, έχουν τοποθετήσει την οικονομία της Ευρωζώνης σε ένα συμπαγές μονοπάτι ανάπτυξης που καθοδηγείται από ενδογενείς δυναμικές και άρα αντιστέκεται περισσότερο σε δυνητική ε, καθυστέρηση της παγκόσμιας ζήτησης ή στέρηση μάλλον της παγκόσμιας ζήτησης. Ταυτόχρονα ο πληθωρισμός φαίνεται να δείχνει ε, σημάδια μιας μόνιμης ανωδικής προσαρμογής προσαρμογής αφού για διάφορα χρόνια έμεινε στάσιμος με, συγκεκριμέ... με, ορισμένες ε, ε, καθοδικές τάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, τα τελευταία, χρόνο παρέμενε, τα τελευταία τρία χρόνια μάλλον παρέμεινε σχετικά σταθερός ο πληθωρισμός, ενώ οι αλλαγές αυτές έχουν ε, καθοδηγηθεί από τις κινήσεις σε πιο ε, κειμενόμενα συστατικά του, όπως οι τιμές της ενέργειας. Σε σχέση τώρα με τις πληροφορίες που έχουμε για τις δυναμικές του πληθωρισμού, οι περισσότερες έχουν μείνει σταθερές. Το τρόφιμα ήταν στο 1% τον Ιανουάριο και αυξήθηκε στο 1,2% από τον Απρίλιο του 2017. Τώρα θα εστιάσω στους τομείς, στους παράγοντες μάλλον, σε σχέση με αυτή την, ε, τον μέτρο πληθωρισμό από μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη μάλλον προοπτική. Αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε δει θετική οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια που στηρίζει ε, μία σταθερή απορρόφηση της οικονομικής ύφεσης. Αυτό προκάλεσε το ερώτημα για το ποιοι παράγοντες κυκλικοί ή διαρθωτικοί μπορεί να έπαιξαν ρόλο στην σχέση μεγέθυνσης με πληθωρισμό. Καταλήξαμε ότι μέσω μιας ανάλυσης του Eurosystem ότι υπάρχουν κάποιοι κυκλικοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς ε, εξελίσσεται ο πληθωρισμός. Είναι ωστόσο το προσωρινή φύση και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το πληθωρισμό μέσω πρόθεσμα, ενώ ακόμα κι αν επηρεάσουν ή και όντως επηρεάζουν το ταχύτητα του της προσαρμογής και του πληθωρισμού. Επιπλέον, δεδομένες της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά την μέτρηση της οικονομικής ύφησης, τα δύο ποσά θα πρέπει να μετρηθούν, πράγμα το οποίο μπορεί να καθυστερήσει την πίεση των τιμών. Αυτό είναι ορατό στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα, όπου η αύξηση των μισθών είναι πολύ μικρή παρά το ότι έχουν αυξηθεί οι θέσεις επασχόλησης. Όμως αυτά όλα θα ξεπεραστούν καθώς θα ε, συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη και θα μειωθεί περαιτέρω η ανεργία. Μάλιστα η αύξηση των μισθών στην Ευρωζώνη τελευταία έχει αυξηθεί και η αγορά εργασίας αναμένεται να βελτιωθεί περισσότερο. Από τη διαστατική πτυχή η παγκοσμιοποίηση μπορεί να έχει μειώσει την ανταπόκριση ε, του πληθωρισμού στις ε, εσωτερικές κυκλικές εθίκες, όμως ε, οι εμπειρίες μας από την Ευρωζώνη δεν είναι ξεκάθαρες για το κατά πόσο δηλαδή οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν αλλαγές στη συμπεριφορά που μπορεί να οφείλονται σε, αλλαγή, σε τεχνολογικές εξελίξεις, όπως ας πούμε η διαφάνεια των τιμών. Ακόμα όμως και αν αυτοί οι παράγοντες είναι κάπως πιο ομόνιμοι, και επίμονοι δεν θα κανονικά δεν θα επηρεάζουν μόνιμα τον πληθωρισμό. Εν γέννη, η ανάλυση δείχνει πως η σχέση ανάμεσα στην μεγέθυνση και στον πληθωρισμό παραμένει ανέπαφη, ακόμα και αν προσωρινώς είχε αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, στο βαθμό που ε, ο βαθμός προσαρμογής του πληθωρισμού προς τους δικούς μας στόχους έχει επηρεαστεί. Τώρα για το μέλλον προβλέπουμε πως ε, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται και σταδιακά μάλλον να προσαρμόζεται προς τα πάνω, στηριζόμενος από τα δικά μας νομισματικά μέτρα Έχουμε λοιπόν ε, πρόσφατα ε, δοκιμάσει ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ενωματικές ισοτιμίες, πράγμα που πρέπει να παρακολουθούμε στενά. Ενώ λοιπόν ε, αυτή η καλή περίοδος στην οικονομία της Ευρωζώνης ε, μας έχει τονώσει την εμπιστοσύνη. Χρειάζεται ακόμα υπομονή και επιμονή όσον αφορά την νομισματική μας πολιτική, ώστε ο πληθωρισμός να μένει κάτω και κοντά στο 2%. Μάλιστα η εξέλιξη του πληθωρισμού καθορίζεται από έναν μεγάλο βαθμό νομισματικής ε, ε, προσαρμογής που παρέχουν τα δικά μας νομισματικά μέτρα. Σημαντικό στόκ ε, μετοχών, επενδύσεις, καθώς και η καθοδήγηση όσον αφορά τα επιτόκια. Τώρα, όσον αφορά το κεντρικό εκαθαριστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και τις δομές ε, εντό της αγοράς που εσείς επιλέξατε ως ε, τίτλο για τη σημερινή ακρόαση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα επίσης. Θα ήθελα να σας θυμίσω το σημαντικό ρόλο που παίζουν ε, οι κεντρικοί ε, CCPs στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενώ ε, ε, διαμεσολαβούν σε ένα δίκτυο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μειώνουν το, το κίνδυνο και αυξάνουν την διαφάνεια της αγοράς. Ωστόσο, υπό συνθήκες κρίσης, η ρήξη των καθαριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις δυνατότητές μας να διεξάγουμε να διεξάγουμε τις νομισματικές μας πολιτικές. Για παράδειγμα, μπορεί να σημάνει ιδιαίτερη ένταση ε, για τη χρήση ρευστότητας για τους χρήστες CCP. Και αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη και ευνίδια ανάγκη για περαιτέρω πόρους ε, σε ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στην αγορά. Αυτό λοιπόν μπορεί να εμποδίσει τα συνήθη, ε, τις συνήθειες διόδους ε, νομισματικής πολιτικής. Αυτά είναι δύο παραδείγματα ε, για τις επιχειρήσεις ανάμεσα στο CCP και την ε, μεταφορά της νομισματικής πολιτικής. Η εισαγωγή ε, υποχρεωτικών ε, απαιτήσεων εκαθάρισης έχει καταστήσει την αγορά πιο διαφανή και αυτό χάρη στην όθηση και στην πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την σύσταση του EMR. Βέβαια, αυτό σημαίνει πως τα CCPs ε, έχουν γίνει πιο συστημικά. Η απόφαση δε του Ηνωμένου Βασιλείου για να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι υπό την τρέχουσα νομοθετικό καθεστώς αρκετά CCPs που ε, καθαρίζουν ε, μεγάλο όγκο ε, συναλλαγών θα λειτουργούν εκτός του πλαισίου των ευρωπαϊκών κανονισμών και των ασφαλιστικών δικλείδων που παρέχονται από αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση της Κομισιόν MER2 που συζητάτε αυτή τη στιγμή την Επιτροπή σας είναι μια ευπρόσδεκτη και απαραίτητη πρωτοβουλία. Το υφιστάμενο καθεστώς ποτέ δεν είχε στόχο να αντιμετωπίσει μεγάλο κλίμακα ε, συναλλαγών σε ευρώ που θα γίνονταν εκτός της Ένωσης. Η πρόταση λοιπόν MR2 θα επιτρέπει στις αρχές να επιπτεύουν αυτόματα συστημικά σημαντικές τρίτες χώρες και τα CCP τους επί τη βάση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών απαιτήσεων χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα. Η πρόταση προβλέπει ευξημένο ε, ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας Έκδοσης και έτσι τονίζει τις τις στενούς δεσμούς ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και την ε, τράπεζα έκδοσης σύσταση για τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6 τον περασμένο Ιούνιο ομόφωνα ήταν πολύ σημαντική και το ε, Δικαστήριο του Λουξεμβούργου στην απόφαση του του 2015 είπε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τροποποιήσει το 22 εάν θεωρηθεί ότι το να έχει την αρμοδιότητα ρύθμιση των ΣΥΣΥΠΗΣ είναι απαραίτητο για την ε, εκπόνηση των ε, καθηκόντων τη υπό τι συνθήκε τη Ένωση. Για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ε, διεκπαιρεώσουμε τα καθήκοντα που μας αναθέτει το MR2, είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις αρμοδιότητες υπό τις συνθήκες και άρα η αναθεώρηση του 22 είναι απαραίτητο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυτή η φάση είναι απαραίτητο να εξοπλιστούμε με τα απαραίτητα μέσα απέναντι στο CCP, ιδιαίτερα για περίπτωση κρίσης. Να εξασφαλίσουμε δε ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους σε ένα περιορισμένο αριθμό τομέων που είναι σημαντική για την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και στην ε, κίνηση προς τις ε, συναλλαγές και τα συστήματα πληρωμών που είναι σημαντικά για να διατηρηθεί η σταθερότητα των τιμών όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Έχουμε λοιπόν ρυθμίσεις ρευστότητας, ε, ρυθμίσεις ε, περιθώρια και ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Να τονίσω ότι τέτοια μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο αν υπάρχει πραγματική απειλή στην άσκηση της συνομισματική μας πολιτική και σίγουρα δεν θα επηρεάσουν τις ε, αρμοδιότητες και τις δυνατότητες των CCP η ΕΚΤΕ θα ενεργήσει μόνο εντός των αρμοδιοτήτων της, δηλαδή να διατυπώνει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική της Ένωσης. Οποιαδήποτε δε μέτρα που θα ληφθούν από αυτές τις βάσεις θα πρέπει να είναι αναλογικά και πλήρως αιτιολογημένα από την ανάγκη της ε, ε, εφαρμογή και τη υλοποίηση του καθήκοντό μα, δηλαδή τη νομισματική πολιτικής. Το καθεστώ εφαρμογή για τις χώρε εκτό Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εξαρτάται όσο γίνεται περισσότερο από τη συνεργασία ε, με τις τοπικέ αρχές. Επίσης να τονίσω πόσο σημαντική είναι η ολοκλήρωση ε, κομματιών κλειδιών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όπως το MR2 πριν από το Brexit ώστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε, ε, για κάθε ενδεχόμενο ακόμα και για το σενάριο που δεν θα ευρεθεί συμφωνία γιατί διαφορετικά οι επόπτες δεν θα έχουν τις δυνατότητες, τη δυνατότητα να χειριστούν τους κινδύνους ε, ε, που μπορεί να σημαίνει η CCP να λειτουργούν εκτός ε, της νομοθεσίας της Ένωσης. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το συστημική διασυνοριακή επίπτωση του κεντρικού εκαθαριστικού μηχανισμού εντός της Ένωσης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυξημένη εποπτική σύγκληση εντός της Ένωσης ώστε να συμβάλλουμε στην ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς και σε ισότιμο πεδίο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί στην επιδίωξη και επίτευξη των στόχων και κλείνοντας να πω ότι τα μέτρα νομισματικής πολιτικής είχαν αυτό ωφέλη για την ε, οικονομία της Ευρωζώνης, αλλά χρειάζονται περαιτέρω πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να περιοριστεί τούν οι αδυναμίες, να ενισχυθεί η αντοχή σε περίπτωση κρίσης και να αυξηθεί το δυναμικό ανάπτυξης. Μόνο φιλόδοξες πολιτικές θα δώσουν συγκεκριμένο ωφέλη στους λαούς της Ευρώπης. Επίσης αυτό μας λέει και η κοινή μας ιστορία. Φέτος ε, ορτάζεται η 25η επέτειος της ενιαίας αγοράς και της συνθήκης του Μάστριχτ ε, και της έναξης ισχύως τους. Αυτές ήταν πολύ τολμηρές αποφάσεις που μας ευνοούν και μας ωφελούν ακόμα και σήμερα. Αγαθά, άνθρωποι, υπηρεσίες και κεφάλαια μπορούν να μετακινούνται ελεύθεροι και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εξασφαλίζει ότι οι κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Με τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Περοχωρήσαμε ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος και σε αυτό το πνεύμα προσβλέπω τους επόμενους μήνες τις συζητήσεις που θα έχουμε για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Εκτιμώ την επιμονή σας και τις ανησυχίε ανησυχίες που αναφέρατε για την οικονομική και κοινωνική πολιτική και για την αφορά που κάνατε και στο νομοθετικό μας έργο. Και το 2022 ε, έχουμε δεσμευτεί λοιπόν να ολοκληρώσουμε το έργο μας μέχρι το τέλος του έτους για τους λόγους που τον είσατε. Τώρα, να, περιοριστώ, να περιοριστούμε στον και να πω ότι στο τέλειο της Ολομέλης στο Στρασβούργο είπατε στην πρότασή σας να επισκεφτείτε τα κράτη-μέλη σε σημαντικές ε, κινήσεις και καταθέσεις ε, πολυεθνικών σε ευρωπαϊκές τράπεζες. 15% ε, τράπεζες της Ευρωπαϊκής προς, το ΕΠΑ, προς τις για να κερδίσουν ακριβώς αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και δεύτερο ερώτημα σε ό,τι η ΕΚΤ έχει λάβει υπόψη τη διάσταση της προστασίας των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την οδηγία που δίνει στις τράπεζες με μη ξεπεριμετωμένα τράνια. Μήπως το... Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Η φορολογική μεταρρύθμιση στη ΣΥΠΑ αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή πολιτική στο δίκαιο και το βλέπουμε ήδη. Είναι μεγάλο εκροές αυτή η μεταρρύθμιση της πολιτικής, ο επαναπατρισμός αυτών των μεγάλων ομίλων και των μεγάλων ποσών που λαμβάνουν οι εταιρείε αυτές συνδέεται ως στοιχεία για την αγορά. Άρα παρατηρούνται αυτές οι ροές. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε μακροπρόθεσμα ποιες θα είναι οι συνέπειες και τα αποτελέσματα. Δίκος αντίκτυπος σίγουρα θα υπάρξει, αλλά δεν ξέρουμε σε τι έκταση από την Αμερική προς την Ευρώπη. Για το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, δεν... Πρόεδρε. Συχνά. Δηλώνετε και την ελπίδα και την πρόθεση προκειμένου Οικονομική και Νομισματική Ένωση περιστάσει. αναφέρεται την ανάγκη να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Ένωση και να την ε, κάνουμε να προχωρήσει. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό θα ήθελα να σας ε, ζητήσω τι πιστεύετε για την τρεχούσα κατάσταση, για την ε, αντιρισμό των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιστεύετε ότι η συζήτηση όπως διεξαγάγεται στους κόλπους του Συμβουλίου μετά την συναντήση κυκλισμένων των θύρων ε, που, ε, συμβιβασμού που πρέπει να υπάρξει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι πιστεύετε σε ό,τι αφορά τη σύσταση και τη σύνθεση εξαρτησία των θεσμικών οργάνων η οποία θα πρέπει να υπάρχει και την οποία διακρίνεται. Αυτό ρυθμίζεται από τις συνθήκες για τη λειτουργία του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 283. Και για την έκθεση στο άρθρο 11, ο Αντιπρόεδρος τα αποσύνθεση της ΕΚΟΦΗΝ, στην επίσημη σύσταση της, ακολουθώντας τις διάφορες διαδικασίες που θετική έχει δηλώσει θετική στάση έναντι του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Αυτό που πετύχει ως τώρα και σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε το στόχο αυτό. Έχω και μισό λεπτό ακόμα, λέει η κυρία Περές. Δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου πλήρω. Δεν ήθελα να μου διαβάσετε τα άρθρα της συνθήκης, να μας ερμηνεύσετε θα θέλαμε σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 283. Η τράπεζα στους κόλπους του Συμβουλίου Κοιτάξτε. Αυτό δεν μπορώ να το συζητήσω εγώ στην παρούσα φάση των υποψήφιων δηλαδή που πρότεινε η ΕΚΟΦ. Να σας πω την εξαρτησία. από τη συνθήκη. Αυτό, ξέρετε, είναι πέρα από τις προσωπικές ε, προτιμήσεις και ο υποψήφιος ε, θα εκτιμηθεί βάσει των κριτηρίων αυτών. Όπως είπατε, λοιπόν, η ΕΚΤΕ θα γνωμοδοτήσει σύντομα. Πότε είπατε, 20... 21 Μαρτίου αναφέρατε ως ημερομηνία, όχι. Νωρίτερα, στις 8 Μαρτίου θα έχουμε την τοποθέτηση της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο, σε ό,τι αφορά το κύριο του και την ελληνικό πλαίσιο. Είναι η πιο σημαντική ασπίδα έναντι των πολιτικών επιρροών σας. Ευχαριστώ, uh, Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντράγκη. Θα ήθελα να εστιάσω στο πρώτο τμήμα της ε, ομιλίας σας. Είπατε για στενή παρακολούθηση. Σκοπεύετε να συμπεριλαμβάνετε στου στους δείκτες μέτρησής σας και τις ε, και τις, ε, και τις τιμές ε, άλλων προϊόντων σκέφτεστε να, να, να συμπεριλάβετε και τις ε, τιμές ε, της ιδιοκατοίκησης στον, στον δίκτυ. Επίσης αναφέρθηκε πρόσφατα ότι η Eurostat σκέφτεται να εισάγει και, τις, ε, και, το, και την ιδιοκατοίκηση για τον υπολογισμό του εναρμονισμένου ε, δίκτυ τιμών καταναλωτή. Θα μπορούσατε ίσως κατά, κατά μια δεύτερη επιλογή να χρησιμοποιήσετε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις ε, ε, τιμές αυτών και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί φούσκα στην αγορά. Ευχαριστώ. Ναι, εξετάζουμε τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, αλλά γνωρίζετε ότι είναι σημαντική πληροφορία. Ο βασικός μας στόχος όμως είναι ο, πληθωρ, πληθωρισμός μάλλον του εναρμοσμένου δίκτυ τιμών καταναλωτή να κινείται ε, κάτω και κοντά στο 2%. Ε, είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι η εστίαση στις ε, τιμές καταναλωτή είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, είναι σημαντικές οι τιμές αυτές ακριβώς γιατί επηρεάζονται και με, ε, επηρεάζουν και τις 3 στα 4 λεπτά. Δύο όμως έχω καταναλώσει κύριε Πρόεδρε. Οπότε καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι δεν θα λαμβάνετε υπόψη τις 3 στα 4 λεπτά. Δύο όμως έχω καταναλώσει κύριε Πρόεδρε. Οπότε καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι δεν θα λαμβάνετε υπόψη τη δεύτερη, από το δεύτερο σκέλος σας καταλαβαίνω ότι δεν θα συμπεριλαμβάνετε στον δίκτυο όλες τις τιμές περισσοκών στοιχείων. Ε, παρά το γεγονός ότι και, και η χρηματοπιστητική ε, κρίση οφείλεται σε ένα βαθμό στο. Να σας πω τι ακριβώς εννοούσα με την απάντησή μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εξετάσει κανεί του λόγου που οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Πρώτον ήταν η επέκταση τη νομισματική πολιτική. Αλλά υπάρχει και άλλο τρόπο για να το εξετάσουμε το θέμα. Και αυτό είναι η αποδιάρθρωση των, ε, ε, των χρηματοπιστωτικών κανόνων που, είχαν, ε, που είχε προηγηθεί κατά 10 χρόνια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις λοιπόν και υπάρχουν αντίστοιχα υποστηρικτές της μίας ή της άλλης εξήγησης. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή που έχουμε μια επεκτατική νομοσματική πολιτική που αιτιολογείται από την τρέχουσα κατάσταση και από, από, από μία άποψη είναι και απαραίτητη βάση της εντολής μας. Δεδομένως όμως της κατάστασης που έχουμε σήμερα, το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε είναι να υπάρξει μια αποδιάρθρωση ή αποδυνάμωση των ε, κανόνων που έχουν θεσπιστεί. Και εγώ μιλώ όχι μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας το λέω αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Wolf Klintz. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι δύο στόχοι που αναφέρονται διαρκώς. Ε, ε, το λέω αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Wolf Klintz. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι δύο στόχοι που αναφέρονται διαρκώς. Ε, ένα βασικό εμπόδιο είναι το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Πότε πιστεύετε και με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, δηλαδή το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μην υπερβαίνει το 10% στις χώρες αυτές. Δεύτερο ερώτημα. Ένα ε, γερμανικό περιοδικό αναφέρει ότι εσείς ε, ήρθατε αντιμέτωπος με τους υπουργούς ε, υπουργού οικονομικών λέγοντας ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να βγει στις αγορές στο, επόμενο, στο άμεσο μέλλον. Και εδώ το ερώτημα μου είναι πότε μπορείτε, πιστεύετε ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί. Επίσης, πιστεύετε ότι ένα τέταρτο μνημόνιο πρόγραμμα διάσωσης ε, θα ε, απαιτηθεί και πώς θα, ε, τι, τι μορφή θα πάρει. Επίσης, μιλώντας για την αναθεώρηση του ΕΖΑΣ με διάφορους συνομιλητές, μαθαίνω ότι το ESRB δεν ε, επικοινωνεί με ακρίβεια και σαφήνεια τις πολιτικές του. Ε, φαίνεται ότι χρησιμοποιηθεί αλγόριθμους και μοντέλα που δεν είναι εύληπτα από, τους, από που είναι έξω. Πιστεύετε διάστημα. Να σας πω για το τελευταίο που ρωτήσατε αρχικά. Δεν το γνώριζα. Αν όμως ε, είναι έτσι τα πράγματα, εμείς βεβαίως είμαστε ε, βελτιωθεί η επικοινωνία μας. Δεύτερο, για το δεύτερο ερώτημά σας, σχετίζεται με τη δημιουργία, ε, θέλω να, να, να, μετριαστούν όσο γίνεται η κίνδυνη κίνδυνοι Άρα η μείωση του κινδύνου, κατά τη γνώμη της ΕΚΤ, θα πρέπει να συμβαδίζει με, την, με τον καταμερισμό, τον επιμερισμό του κινδύνου. Τμήμα της μείωσης του κινδύνου φυσικά αφορά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά όχι μόνο. Ε, συνδέεται και με τα περιουσιακά στοιχεία επίπεδο 2 ε, και 3 που εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτή είναι η κληρονομιά άλλωστε της χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και της μεγάλης ύφεση. Όλα θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν και τα δύο. Αν θέλουμε Είτε θέλουμε ποσοτικούς στόχους είτε όχι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουν οι επόπτες. Γενικά οι επόπτες δεν θέλουν να τους λένε άλλοι ποιοι είναι οι αριθμητικοί στόχοι που πρέπει να εφαρμοστεί σε, σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης, γιατί θέλουν να διατηρούν τη ε, διακριτική ευχέρεια να εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Φυσικά ε, χρειάζονται εκθέσεις προόδου ποιοτικού χαρακτήρα ε, και νομίζω ότι έχετε δίκιο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τέλος, για την Ελλάδα. Όχι. Νομίζω ότι αναφερθήκατε. Υπήρχε μια παρουσίαση και αφορούσε και τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ε, ανάγκη μείωσής τους μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και να σημειωθεί πρόοδο. Και να σα πω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά υπάρχουν ακόμα, ε, ούτε συζητήσαμε φυσικά κάποιο περαιτέρω πρόγραμμα και προφανώ και δεν είναι δουλειά του Προέδρου τη ΕΚΤ να πει κάτι τέτοιο. Εξαρτάται από τον ESM. Ο κύριος ε, ε, Τσακαλώτο είπε στην ουσία το ίδιο. Ότι το θέμα πήρε υπερβολικά μεγάλε διαστάσει Που είστε για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας παρών, και χαίρομαι ιδιαίτερα αλλά και γιατί περιγράψατε με τα ίδια ακριβώς λόγια με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο αυτό που ορισμένα μέσα ενημέρωση στην πατρίδα μου την Ελλάδα το εμφάνισαν ως ένα πολύ μεγάλο καυγά, μια πολύ μεγάλη διαφωνία ανάμεσα στο Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου και ο κύριος Σεντένο και ο κύριος Μοσκοβισή και ο κύριος Ρέκλινγκ επιβεβαιώνουν ότι με τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί από τις ελληνικές αρχές βαδίζουμε προς την έξοδο της Ελλάδας από, το, από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε επίσης στο ίδιο μήκο κύματο την αναβάθμιση με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετέχει στο κουαρτέτο των θεσμών να μας πείτε και τη δική σας εκτίμηση για αυτές τις προοπτικές. Είστε στο ίδιο μήκο κύματο με τους κυρίους Σεντένο, Μοσκοβισή, Ρέκλινγκ με τα συμπεράσματα των οίκων αξιολόγηση ότι με την πρόοδοξη εκτίμηση ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι. Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξος. Όλες οι συμφωνηθέν συμφωνηθήσεις δράσεις έχουν εφαρμοστεί. Οχι ότι ε, θα υπάρχει συνεχής, απρόσκοπτη ε, υλοποίηση των πληστηριασμών χωρίς γεωγραφικούς ε, αποκλεισμούς και περισσότερο κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, έχω ένα ερώτημα σχετικά με την αποτυχία της τράπεζας ABLV. Αναφέρθηκε ότι η ABLV έλαβε δύο φορές ε, χρηματοδότηση και την Τετάρτη πριν την Παρασκευή και το Σάββατο τελικά ε, αποφασιστεί η χρεοκοπία της. γιατί λοιπόν ε, δόθηκε αυτό το πρώτο ELA όταν ήδη είχε ε, μπει η κατάσταση σε καθεστώς παγώματος. Δεύτερον, για να χρεοκοπήσει. Και είναι, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο σα την Τετάρτη και την Παρασκευή το βράδυ. Και τι τελικά, ποιο τελικά είναι το δίδαγμα σχετικά με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ELA και την εποπτεία των τραπεζών. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σχολιάσω ε, λεπτομέρειες ε, των δραστηριοτήτων το ELA πέραν των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι ίδιες οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Άλλωστε e, το ELA δίνεται από τις ίδιες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και αντίρρηση μπορεί η ΕΚΤ να εκφράσει μόνο όταν υπάρχει πλήγμα για, την, ε, για τους στόχους της νομισματικής μας πολιτικής. Και οι πληροφορίες ε, που δίνουμε εμείς καλύπτονται από τη συμφωνία ELA. Η πρόληψη λοιπόν νομιμοποίησης παράνομων ε, δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντική, αλλά η διάταξη του ELA καλύπτει συγκεκριμένη κεφαλαιακή ανάγκη της τράπεζας ε, περισσότερα, περισσότερες πληροφορίες δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω. Uh, uh, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση αυτή την οποία και αναμέναμε. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω το εξή. Ε. Μήπως πιστεύετε ότι τέτοιες περιπτώσεις ε, αμφισβητήσιμη χρήσης ή λέει ουσιαστικά βλάπτουν την αξιοπιστία του συνολικού συστήματος και άρα οι πολιτικές ΕΛΑ θα έπρεπε να τροποποιηθούν. Και μια τελευταία ερώτηση για τις συστάσεις ε, του διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά και τους G30. Θα την λάβετε υπόψη τη σύσταση αυτή της διαμεσολαβητρίας. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την τελευταία σας ερώτηση, σημειώνουμε ασφαλώς την απάντηση και την ε, επιστολή της ε, διαμεσολαβητριάς και θα της δώσουμε απάντηση στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο. Μέσα Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο τώρα. Συμφωνώ μαζί σας. Ε, η πολιτική λέει θα πρέπει να αλλάξει. Και εγώ σε διάφορες περιπτώσεις έχω διακηρύξει την ε, κεντρικό, κεντρική διαμορφώση του ELA. Αυτό αποτελεί, αν θέλετε, ένα υπόλοιμα παλαιότερων καιρών. Θα πρέπει όμως να υπάρξει συμφωνία όλων των χωρών, όλων των ελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου προκειμένου να γίνει η αλλαγή αυτή για να εγκαταλείψουμε αυτό το υπόλοιμα εθνική κυριαρχία στην νομισματική πολιτική, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτά ήθελα να πω στην παρούσα φάση. Σας ευχαριστώ, Μάρκο Βάλλη. Eh, ευχαριστώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό που, όπως, που είπατε, ε, σε σχέση με αυτό που είπατε πέρα από το 2018 ως ημερομηνία καταληκτική αν δεν, τηρηθούν, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Δεν θέλω μια κοπία λόγω τέτοιων περιστάσεων. Ε, σκέφτεστε να φτιάξετε ασφαλή ομόλογα, να είναι ένα μέσο... Έπειτα, η, ότι τα δεύτερο και τρίτο επίπεδου καλύπτεται από τα κεφάλαια των τρισσότερων για να αποφύγουμε συστημικούς κινδύνους. Νέες ε, παρατάσεις ε, ποσοτικής χαλάρωσης δεν έχουν συζητηθεί. Αυτό που δεν είμαστε πεπισμένοι πως ο πληθωρισμός προχωρά προς το στόχο μας, αλλά πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και επίμονοι, διότι για τους επόμενους μήνες. Η πολιτική παρακολούθηση τώρα ε, και η αποτελεσματικότητα αυτής οφείλεται σε συνδυασμό διαφόρων. Επενδύει τα ομόλογα που οριμάζουν για μια μακρά χρονική περίοδο μετά από το πρόγραμμα Net Asset Purchase. Τώρα, δεύτερο σα ερώτημα αφορά την δημοσιονομική σύγκληση και τη δημιουργία ενό ομολόγου το οποίο να είναι ένα ασφαλέ στην Ένωση ώστε οι χώρε να είναι σε θέση να επιβιώσουν καλύτερα στην κρίση. Η αλληλεγγύη έρχεται με την ευθύνη και την υπευθυνότητα στην Ένωση ώστε οι χώρε να είναι σε θέση να επιβιώσουν καλύτερα στην κρίση. Η αλληλεγγύη έρχεται με την ευθύνη για την υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα σημαίνει σύγκληση των οικονομικών πολιτικών, σύγκληση των οικονομικών δομών και σύγκληση προς την καλύτερη πρακτική όσον αφορά τους θεσμούς. Μάλλον αυτό είναι και το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό είδος σύγκλησης δηλαδή. Και η ίδια σύγκληση ε, δημιουργεί την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη ώστε να έχουμε ένα κοινό ασφαλές ε, στοιχείο. Δεύτερο ερώτημα. Βεβαίως πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια είναι, καλύπτουν επαρκώς αυτούς τους κινδύνους και ότι ούτως ή άλλως η ΕΚΤ τώρα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκτίμηση μοντέλων που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τα, τα στοιχεία επίπεδο 2 και 3. Και αυτά θα πρέπει φέτος μάλιστα να ξεκινήσουν. Μάλιστα. Εμείς το συστήναμε Είναι αυτό. Το συστήνει λοιπόν αυτό. Κύριε Κάπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράκη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε παρά τι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Να επικεντρωθώ στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόεδρε Ντράγκη, σας ευχαριστώ που ήρθατε παρά τι δυσκολίε που αντιμετωπίσατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Να επικεντρωθώ στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γνωρίζετε το, την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση των μη ε, εξυπηρετούμενων δανείων. Θετική συνολικά Έχουμε 950 δις ακόμα συνολικά, αλλά είναι καθοδική η τάση. Ο όγκος είναι υψηλός ακόμα, μελών από 0,7 ίσως 40 και κάτι της 100. Για εκδώσατε μία, ένα συμπληρώμα για τις καταφυντέντριες οδηγίες ό,τι αφορά τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε ό,τι αφορά την ποσοτική διάσταση, σε ό,τι αφορά την ε, διάσταση του ρίσκου, για το που παλιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα εκδοθεί ένα κατάλογος για τα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη σύγκληση, έχουμε να πούμε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα, τις εταιρικέ ε, τράπεζες, η Ελλάδα αναφέρθηκε και εδώ στην Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύτηκε μια έκθεση ελέγχου τα μέτρα τα οποία προτείνονται το πρώτο τρίμηνο σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και επίσης η κατάσταση στην Ελλάδα και η κατάσταση στην Ιταλία πώς την εκτιμάτε. Θα ήθελα καταρχάς να πω το εξή Σε ό,τι αφορά τα... την αντιμετώπιση, τη συστηματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτό είναι δεδομένο γιατί επηρεάζουν ε, την λειτουργία των τραπεζών μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Άρα οι τράπεζε με υψηλά NPL, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ε, τελικά βλάπτουν την ε, ανάπτυξη. Δεν δίνουν αρκετά δάνεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την. Πάει πακέτο με την μείωση του επίπεδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και είπατε και στι χώρε που αναφέρατε, αλλά και σε άλλε χώρε έχει μειωθεί ο ρυθμό των δανείων αυτών. Και το επίπεδο των διατάξεων έχει αυξηθεί η φραγκιότητα, η κερδοφορία του τραπεζικού συστήματο. Όλα έχουν βελτιωθεί. Έχουμε τώρα πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κοιτάξουμε το θέμα των δανείων αυτών στον πρώτο πυλώνα. ορίζουμε την πρόταση του επίπεδου για καινούργια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό το οποίο αποκαλείται αυτόματι κανόνες ε, πρώτου πυλώνα. Αυτό όμω είναι διαφορετικό. Το αντέντομ, το παράρτημα που αναφέρατε έχει να κάνει με εποπτικές προσδοκίες αντίθετα με το προσάρτημα αυτό. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν δεσμευτικές προδιαγραφές και θα ισχύσουν αυτόματα σε όλα τα θεσμικά όργανα. Ο επόπτης θα πρέπει να εκτιμήσει το προφίλ κινδύνου και τις ε, συνθήκες που τον καθορίζουν. Αυτό τι σημαίνει ότι αν οι διατάξεις ε, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για το κάθε θεσμικό όργανο έχουν να κάνουν με το θυμίο αυτό, θα πρέπει να μην υπάρχει υπόλοιπο κίνδυνος και θα χρειαστούν ε, μέτρα δεύτερου πυλώνα. Αν δεν ε, επιβεβαιωθούν οι άλλες ε, συνθήκες, τότε θα χρειαστούν τα διατάξει του δεύτερου προσαρτήματος. Άρα ουσιαστικά είναι άλληλο συμπληρωματικά, μάλιστα, η για τους επόπτες σε βάθος χρόνου. Και τώρα, δυστυχώς, θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε τους ομιλητές μας, γιατί στις 5.25 πρέπει να ολοκληρώσουμε. Γιατί έχουμε να επιτελέσουμε και τα καθήκοντά μας που ορίζει η συνθήκη σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο στη θέση του Αντιπρόεδρου του ΕΚΤ. Είναι σπουδαία ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας. Ο ρόλος της ήταν ε, πολύ σημαντικός για την οικονομική ανάκαμψη, αλλά δεν αρκεί μόνο η νομισματική πολιτική για να έχουμε μια ισορροπημένη και μόνιμη οικονομική ανάκαμψη. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς τα κίνητρα τα νομισματικά μπορεί να κινητοποιήσουν αυτήν την ανάκαμψη. Και ένα θέμα ήταν οι συναγωματικέ ισονομίες. Θέλω να ξέρω εσείς τι νομίζετε και ποια πιθανά μέτρα μελετάτε. Τι μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν. Μάλιστα, καλησπέρα σα. Δύο πόρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γνωρίζετε, αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στην έκθεση Μόντι και στην έκθεση τη ΕΚΤΕ που εγκρίθηκε πρόσφατα. Χρειάζεται πολιτική ε, βέβαια πλειοψηφία και είναι αλήθεια ότι η ΕΚΤ έκανε το πολύ. Ο κύριος Φανχέν Η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου την περασμένη εβδομάδα ε, έδωσε τη δική της έκθεση και μια από τις ανησυχίες είναι η εξέλιξη της ε, αγοράς, της κτηριακής αγοράς ε, στην Βελκική αγορά λόγω του βάρους που αυτό αντιπροσωπεύει για τα νοικοκυριά οι τράπεζες δίνουν εξαιρετικά εύκολα λένε δάνεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν 1,5 δις ευρώ buffer ε, και βέβαια όσο μεγαλύτερο είναι το χαρτοφυλάκι τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι και αυτό το ε, μέτρο, το buffer. Εσείς σας ευχαριστώ. Γιάκο Ευχαριστώ. Ζούμε πλήρως την άποψη ότι μια κεντρική τράπεζα πρέπει να συμμετέχει. Το ερώτημα όμως είναι τι αν στο μέλλον το κάνουμε αν, για παράδειγμα, συγχωνεύσουμε την ρύθμιση αυτού του θέματος από τον ΕΣΜΑ λόγων ε, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιους τομείς λοιπόν θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα η ΕΚΤ και σε ποιους τομείς η ΕΣΜΑ ή κάποια άλλη ρυθμιστική αρχή της Ένωσης. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε, πιστεύετε ότι πρέπει η ΕΚΤ να τίθεται επικεφαλής και πού ε, ο ΕΣΜΑ, ο κύριο Κίρτσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. διότι Να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το τεράστιο χρέο μα. Δυστυχώ, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο ήταν αρνητικό σε τήσια βάση για την Ελλάδα και αυτό έγινε για πρώτη φορά από το τέλος του 2016. Η ΕΚΤ έχει αναλύσει την κατάσταση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Πιστεύω ότι οι πληστηρισμοί αυτοί θα αρχίσουν σε κάποιες εβδομάδες, κάτι που είναι ε, θετική εξέλιξη βεβαίως. Ωστόσο δεν πιστεύω ότι μπορεί να ε, εξομαλυθεί η κατάσταση εύκολα γιατί υπάρχουν εξοκοινοβουλευτικές. Άρα ε, πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία Δεύτερον, πιστεύετε ότι θα αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Περιμένουμε η Κομισιόν να εκδώσει ένα σχέδιο δράσης με τις πρωτοβουλίες της και ποιες αρμένους ε, κλάδους που ε, αυξάνουν και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωζώνη. Ε, ενώ μόνο 18 και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας καλέσω να είστε και πιο ανοιχτοί και διαφανείς σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη από του άλλου συναδέλφου. Πρέπει να σταματήσουμε τι ερωτήσει. Ε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντράγκη, αλλά να τον, να τον παρακαλέσω ε, να μα τα πει πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Πρώτο ερώτημα. Αν η νομισματική πολιτική είναι το μόνο ή το βασικό εργαλείο για την ανάκαμψη και για την εξυγίανση ε, της υπάρχουσας ανάπτυξης. Όχι φυσικά και το λέω ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έχετε κουραστεί να με ακούτε να το, να το λέω. Το λέω εδώ και πέντε χρόνια. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν και ανησυχούμε ε, για το ότι αυτές οι διακυμάνσεις μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό και αυστηροποίηση. This is political decision. Πρόκειται περί πολιτικής απόφασης και αν θέλω το οποίο θα αντιστοιχεί σε μερίδιο των καθαρών κερδών που ε, προκύπτουν από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην Ευρωζώνη να, μεταφερθεί, να, να μεταφερθούν τα ποσά αυτά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό είναι νομισματική και υπέρ αυτού του είδους των μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίζονται μη συστημικές καταστάσεις όπου οι ο ΕΣΜΑ είναι ο βασικός ε, ρυθμιστής, επόπτης. Η ΕΚΤ θα πρέπει να παρακολουθεί τον κίνδυνο που θέτουν από τις αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ. Φυσικά σε συντονισμό με την ΕΣΜΑ θα κάνουμε τις ενέργειές μας προκειμένου να μην επαναλαμβάνουμε έργο το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί ε, και να περιοριστούν οι διακοιμάνσεις στις αγορές. Με βάση όμως τον κανονισμό ΕΜΙΡ, η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει τις εξουσίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να προχωρά σε αυτού του είδους ενέργειες και βεβαίως εμείς, ε, και, αλλά και άλλες χώρες. Η συνεχιζόμενη βελτίωση της κατάστασης ωστόσο πρέπει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι για την βιώσιμη ε, ε για τις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εμείς είμαστε βεβαίως συμβαλόμενοι. Η ε, φυσικών καταστροφών μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης της οικονομίας και των αγώνων. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, υποστηρίζουμε τις πολιτικές σχετικές, ωστόσο θεωρούμε ότι... την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Το Μάιο περίπου. Περιμένουμε ακόμα επιβεβαίωση της επίσημης ημερομηνία. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Και θα ήθελα να καλώσω, όπως ξέρετε, το Συμβούλιο ΚΟΦΗΝ αποφάσισε στις 20 Φεβρουαρίου να συστήσει τον Ισπανό Υπουργό Οικονομικών κ. Ντεκίνδος ως αντιπρόεδρο της ΕΚΤ για την αντικατάσταση του κ. Κωνστανση από 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους Συμβούλιο ορίζει τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, τον επιλέγει μεταξύ ατόμων υψηλού επαγγελματικού κύρου σε τραπεζικά ζητήματα μετά από διαβούλευση με το, Ευρω... με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το... Α, την Εκκληστική Επιτροπή της ΕΚΤ. Σήμερα λοιπόν η ακρόαση αυτή εντάσσει του υποψηφίου ένα εκτενές ε, ερωτηματολόγιο το οποίο και απάντησα. Σας ευχαριστώ και θα βρείτε ερωτήσει και για θέματα νομισματικής ένωσης αλλά και για θέματα διαβάνειας ότι η Επιτροπή Οίκων διοργάνωσε και ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων με τους δύο υποψηφίους για τη θέση αυτή. Και τώρα λοιπόν εισερχόμαστε στην επίσημη διαδικασία και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κριτική για να μας κάνει... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να εμφανίζομαι εκ νέου σε αυτήν την Επιτροπή για την επίσημή μου ε, ακρόαση ως υποψήφιος ε, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, θα σας μιλήσω για την πορεία μου, την κοινωνική ευημερία. Θα ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ε, την σημασία του να εμβαθυνθεί και να προωθηθεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, όχι μόνο για την εγγύηση μια σωστή διάδοση τη νομισματική πολιτική, αλλά και για το μέλλον του project του ευρώ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι όρθια από την κρίση και εν μέρει λόγω των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που περάσαμε. Το ε, δικό μας οικονομικό σύστημα υπέφερε από προβλήματα διαφάνειας ε, και για να ξεπεραστούν οι αμφιβολίες αποφασίστηκε να γίνει μια βατομέα. Ε, και έτσι μπορέσαμε να ξεφορτωθούμε και ε, τα διάφορα μη εξυπηρετούμενα ε, δάνεια. Ε, ιδιαίτερα επίσης όσον αφορά την ε, λάθος εμπαρευματοποίηση διαφόρων προϊόντων αλλά όπως των διαφόρων ε, ε, επαγγελματικών κλάδων μπορέσαμε να οριθμίσουμε την κατάσταση και να ρυθμίσουμε και τα θέματα αφαιρεγγιότητας αλλά και την εγγύηση. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαλαν στο να ανακάμψει η Ισπανία η ε, Ισπανία θεωρεί 6 χρόνια η πορεία μου στο δημόσιο τομέα επεκτάθηκε ως ε, Υπουργό Οικονομίας όπου μπόρεσα ε, να συμμετέχω στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής και στην περίοδο κατά την οποία η Ισπανία που κανέναν απολύτως δεσμό. Τώρα θα περάσω στο τμήμα που είναι πιο, το πιο σημαντικό, είναι η νομισματική πολιτική της ΣΕΚΤ. Παρακαλώ επιτρέψατε μου να συνεχίσω στα αγγλικά. Τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε από την εμπειρία ότι η πιο σημαντική συμβολή που μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική είναι η σταθερότητα των τιμών. Και είναι δίκαιο να πούμε ότι η ΕΚΤ επιτυχώς έχει επιτελέσει αυτό το στόχο τα τελευταία, ε, στη διάρκεια των ετών. Η ΕΚΤ ε, ε, πάντοτε αντέδρασε δραστήρια υιοθετώντα μέτρα ώστε να αποφύγει τον υπερβολικό πληθωρισμό. Αυτή η επιτυχία βασίζεται έχει βασιστεί σε μια, ένα απλό αλλά αποτελεσματικό νομισματικό λειτουργικό πλαίσιο και μια νομισματική πολιτική που συμπεριλαμβάνει έναν συγκεκριμένο ορισμό για τη σταθερότητα των τιμών με μια δι δι, ε, δι, διπλή ε, προσέγγιση. Ταυτόχρονα όλα αυτά θα είχαν καταστεί δυνατά χωρίς έχει δείξει πως η ανεξαρτησία είναι κρίσιμη ώστε να διατηρεί μια κεντρική τράπεζα χαμηλά τα επιτόκια ε, μέσω πρόθεσμα. Αυτή η ανεξαρτησία είναι απόλυτα εγγυημένη από τις συνθήκες για την, συγκεκριμένα για την ΕΚΤ όπου θεσπίζεται και το σύστημα το ευρωπαϊκό που συναποτελεί από τις λεπτομέρειες, ε, μάλλον ε, πληροφορίες για την ε, συνεργασία και τις στρατηγικές, ώστε να μπορεί να είναι πάντοτε σταθερός ο πληθωρισμός. Έπειτα μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει διαθεσή της και άρα η ΕΚΤ είναι λογοδοτή στους Ευρωπαίους πολίτες επιδιώκει αυτές τις πολιτικές εντός της Ένωσης. Όπως πριν τρεις εβδομάδες δήλωσε ο πρόεδρος Δράγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σκοπεύουμε, ε, σκοπεύει μάλλον η ΕΚΤΕ να διατηρήσει το 2% ανάπτυξη ε, που έχει τα τελευταία τρία χρόνια διαπιστωθεί στην Ευρώπη. Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις ε, σε σχέση με τις ε, πιθανές παρενέργειες ε, συνεχίζονται ωστόσο και θα το γνωρίζουμε και θα ήθελα να αναφέρω πως αυτές οι ανησυχίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το ότι ένα από τα βασικά αρνητικά της χρηματοπιστωτικής αστάθειας μπορεί να είναι η ρήξη των ε, καναλιών επικοινωνίας ε, και μετάβασης. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί η εποχή. Θα ήθελα να μιλήσω για και να τονίσω μία από τις σημαντικότερες ενέργειες, τη μετάφαση και την διαβίβαση αυτής της πολιτικής από την ΕΚΤ προς τα κράτη. Εξαρτάται τόσο από την δομή όσο και από του κάθε κράτους όσο και από την οικονομική της ε, νομισματικής πολιτικής. Η αποτελεσματική ε, λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ε, είναι ουσιώδους σημασία για να μπορεί να μεταφράζεται σε πράξη η νομισματική μας πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να μπορεί η χρηματοδότηση που λέει ότι εγγυόμαστε τις καταθέσεις όλων των καταθετών ανεξάρτητα από αυτές βρίσκονται. Ε, άλλα μέτρα είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων, η απέτηση της τράπεζας για μια στάνταρ δυνατότητα απορρόφησης ε, απολειών και ζημιά. Η ανάπτυξη των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι ένας άλλος στόχος. Από την άλλη πλευρά, για να υλοποιηθούν και να υλοποιήσει τις ευρωζώνες και θα έχουμε και ένα μηχανισμό που θα ελέγχει τις οικονομικές πολιτικές. Αυτή η τωρινή συγκυρία της ανάπτυξης ε, έναντι στην πρόσφατη οικονομική και οικονομική κρίση. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε ότι αυτή η οικονομική πολιτική, η νομισματική πολιτική είναι παντοδύναμη. Ένα, μια γενική αποστολή, ένα μια εντολή, ώστε να είναι ε, ε, ακόμα πιο κατάλληλη η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και γι' αυτό και είναι τιμή μου που το, συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ε, αποφάσισε να με προτείνει προς όφελος και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Κύριος Brian Hayes, πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ. Κύριε Κουίντους, σας καλωσορίζω άλλη μια φορά εδώ στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που παίζουμε εμείς ως μέλη της ΕΚΟΝ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διάλογό μας με την ΕΚΤ. Είδατε ότι είχαμε μαζί μας σήμερα νωρίτερα τον πρόεδρο Ντράγκη. Αυτό είναι μια μόνιμη διαδικασία, καθώς και η έκθεση που συντάσσουμε ετησίως και τις τακτικές ερωτήσεις που απευθύνουμε στην ΕΚΤ ε, μέσω του Προέδρου μας ε, Γκουαλτιέρη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρετε πώς μπορούμε να, να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να έρθουμε σε ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία με την ΕΚΤ δεδομένου του ρόλου που ε, προτείνετε να αναλάβετε εσείς ως Αντιπροέδρου το λέω αυτό διότι ο πρόεδρος Ντράγκη πολύ συχνά αναφέρεται στην λογοδοσία ε, ε, και, την, ε, το διάλογο μεταξύ των Ευρωβουλευτών και, των, και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εσείς στα μελλοντικά σας καθήκοντα πιστεύετε ότι θα έχετε κάτι συγκεκριμένο να, προσ, να, να κομίσετε ως προς αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τον ρόλο των μέτρων για το 2% ε, και την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, σας ανησυχεί το γεγονός ε, ε, ε, ε της συν, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου ευρώ που έχει μειωθεί ε, πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει τον, ε, την επίτευξη του στόχου περί 2% πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ε, στα καθήκοντά μου Υπουργού ε, στην Ισπανία επισκέφτηκα το κάθε δημόσιο εξωματιούχο γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ζωτική σημασία ε, στοιχεία προκειμένου να ενισχύεται και να βελτιώνεται ο διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι ε, στο βαθμό του, του δυνατού θα έρχομαι σε διάλογο έχω να επιδείξω ένα ιστορικό, πολύ θετικό Ω προ τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Και αυτό ακριβώ είναι το, η άλλη... Ήταν θετική και νομίζω ότι λάβαμε σωστέ αποφάσει. Τώρα βρισκόμαστε σε φάση ανάκαμψη. άρα θεωρώ ότι ήταν θετική η σύμβολη του Eurogroup και η Ευρωζώνη αναπτύσσεται πιο ταχαίω σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Αυτό ήταν ασύλληπτο μόλι πριν από δύο-τρία χρόνια. Προφανώ. πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν, λοιπόν, τον οποίο και υποστήριζα. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι θα συνεχίσει το Eurogroup να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την περαιτέρω εμβάθυνση τη νομισματική ε, ενοποίηση. και το πιστεύω. Ναι, θα απαντήσετε και τι υπόλοιπε ερωτήσει, με. Ναι, κοιτάξτε, δεν ε, το, το μέγεθο του ισολογισμού τη ΕΚΤ. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό τη ΕΚΤ, αυτό είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων που προκύπτουν από το... Ως τώρα προσέξη της ΕΚΤ ήταν σωστή και είμαι βεβαίως ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη σωστή νομισματική πολιτική. Ευχαριστώ. Και η Σουίμπορν. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε Υπουργέ και τις εκπροσώπηση των δύο φίλων ε, στην ΕΚΤ. Είναι ένα θέμα που μας ε, συγκινεί γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καλή ισορροπία. Εσείς δεν μπορείτε να ολοκληρώσει τους κανόνες για την, το ευρώ. Μέχρι το 2019. Κοιτάμε λοιπόν το τι γίνεται στα πλαίσια της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Δήλωσε επίσης ότι η ΕΚΤ σε καιρό κρίσης θα χρειαστεί να την δράση Ευχαριστώ πολύ. Τρεμόζα. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο και καλή επιτυχία σας εύχομαι από πλευράς ομάδας μου ε, σε αυτή την υποψηφιότητα της Αντιπροεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά πρώτα κάτι για την ε, εσωτερική τοπική ισπανική πολιτική. Εσεί ε, είπατε ότι είστε υπουργό Οικονομίας και πόσο θεωρείτε ότι είναι ανεξάρτητη η ΕΚΤ και μέχρι πότε θα ισχύει. Θα ήθελα να μας δώσετε τη δική σας γνώμη τώρα για την, για την ε, νομισματική πολιτική. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το Fed, η ΦΕΔ ανεβάζει τα επιτόκια και προετοιμάζει για την επόμενη ύφεση κερδίζει χώρο για μελλοντικέ ενέργειες. Γιατί η ΕΚΤ εξακολουθεί να αυξάνει το ισοζύγιο και διατηρεί στο μηδέν τα επιτόκια. Πιστεύετε πως η ΕΚΤ έχει αργήσει να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα σχετικά με την νομισματική πολιτική και έπειτα σε ποιο επίπεδο νομίζετε και πότε θα πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια στην Ένωση και έπειτα ποιε συγκεκριμένε πολιτικέ θα, σκέφτεστε, θα, σκεφτόσασταν για να μειώσετε ε, το ισοζύγιο της ΕΚΤ. Ναι. Ε, Σήμερα είπε ο Πρωθυπουργό ότι τι επόμενε μέρε εγώ δεν θα είμαι πια Υπουργό Οικονομία και φυσικά είμαι στη διάθεση του, όπω είπε και ο ίδιο, τι επόμενε μέρε. Για τι άλλε ερωτήσει που αναφέρατε σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική, καταρχά, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η θέση στον επιχειρηματικό κύκλο τη Ευρώπη δεν είναι ακριβώ η ίδια με αυτή τον είπα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η θέση στον επιχειρηματικό κύκλο της Ευρώπης δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτή τον ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη και φυσικά είναι πολύ χαμηλότερο και το ποσοστό ανεργία. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό το γεγονός ότι ομοσπονδιακό, αποθεματικό, μάλλον η, το, Κεντρική Τράπεζα στην Αμερική έχει αυξήσει τα επιτόκια για να μειώσει και τον ισολογισμό σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό, τον επιχειρηματικό κύκλο. Δεν νομίζω ότι υστερεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση για την νομισματική πολιτική, αλλά διαφορετικέ διαφορετικές καταστάσεις πολύ απλά. Αν μου επιτρέπετε ωστόσο να διευκρινίσω το εξή του χρόνου, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ πιστεύω ότι θα συγκλίνει προς αυτό που ε, βλέπουμε ότι διαμορφώνει ως πολιτική η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, νομίζω ότι είναι σαφής η πολιτική της ΕΚΤ. Μόλις τον ισολογισμό θα αποτελέσει συνέπεια του προγραμματός αγοράς ομολόγων. Ξεκινήσαμε με 80 δις για την αγορά ομολόγων και τώρα είμαστε στα 30 ανά μήνα. Το μύριο ώρες απασχόλησης χάθηκαν. Οι ερευνητέ μας και οι νέοι μας φεύγουν από την Ισπανία. Και μάλιστα Το μύριο ώρες απασχόλησης χάθηκαν. Οι ερευνητέ μας και οι νέοι μας φεύγουν από την Ισπανία. Και μάλιστα... Τώρα εσείς μας παρουσιάζετε αυτά σας τα διαπιστευτήρια και λέτε ότι η ρευστότητα θα μειώσει το δημόσιο χρέο. Ναι, κλείνω, κλείνω. Εμείς θα σας καταψηφίσουμε κύριε Τεγκίντος. Κοιτάξτε, δεν, δεν είναι αυτή η εξήγηση ψήφου. Εμείς θα σας καταψηφίσουμε. Εσείς είπατε διάφορα σχόλια που νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Πρώτον, αλλαγή στην οικονομία της Ισπανίας. Υπήρξε αλλαγή στην οικονομία εδώ και τρία χρόνια αναπτύσσεται πάνω από 3%. Έχουμε μισό εκατομμύριο θέσει απασχόληση που δημιουργήθηκαν. Ναι, μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, όμω ήδη είναι διαφορετική κατάσταση από αυτήν που είχαμε πριν από 5-6 χρόνια. Και είναι κάτι που κάθε αναλυτής οικονομικός το δέχεται. ούτε η αύξηση των πιστώσεων, ούτε η φούσκα ε, των ε, ε, κτηρίων είναι αυτή η οποία μας δημιούργησε την κρίση. Είχαμε πάντως πολύ χειρότερη κατάσταση προηγουμένως. Τώρα έχουμε και δημιουργήσαμε 40, 40 δις που ήταν το πρόγραμμα διάσωσης και να επαναλάβω ότι συνέπειες τις βλέπουμε. Είχαμε ένα σύστημα δημοσιονομικό σίγουρα ελαττωματικό. Σήμερα οι οικογένειες και οι ισπανικές ε, εταιρείε πληρώνουν επιτόκια παρόμοια με αυτά των ε, Εμείς ε, δεχθήκαμε κατηγορίες ότι δεν σας στηρίζουμε παρότι είστε Ισπανός υποψήφιος. Εμείς θέλαμε να υποστηρίξουμε τον κύριο Κάμπας ε, που είχε και περισσότερες ψήφους ε, αρχικά. Τώρα βέβαια αυτό ήταν για το Eurogroup, τώρα θέλετε να καλύψετε τη θέση του Αντιπροέδρου στην ΕΚΤ. Έχετε όμως ένα πολύ επικίνδυνο παρελθόν. Τι θα γινόταν με το άρθρο 7 του καθεστώτος ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και αυτό είπατε αυτό στη δική σας ε, ε, εισήγηση και είπατε ότι μάλιστα αυτό το θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων. Επίσης, εσείς μυρίσατε, εσείς ήδη έχετε δουλέψει στο ταμιευτήριο, ε, το ιδιωτικό, μετά σώσατε ως υπουργό στην ίδια τράπεζα, με πολλά εκατομμύρια τράπεζα, γιατί μπέμεν το ίδιο, εσείς ήσασταν ανεξάρτητος σύμβουλος και ήσασταν και μέλος μετά της εποπτείας και του ελέγχου της ίδιας τράπεζας, την οποία διασώσατε με... Ε, ε, σε συμφερόντων είπατε ότι ποτέ δεν θέλετε να απειλήσετε τέτοιες ε, τις τράπεζες αυτές και παρόλα αυτά στο ίδιο σας το βιβλίο ε, το οποίο εσείς γράψατε, είπατε για αυτές τις τέσσερις ε, διαμεσολαβήσατε ή όχι. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Εγώ νομίζω πως ναι, διαμεσολαβήσατε. Ε, και τι εγγύησεις μας δίνετε ότι τώρα δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω πρώτα απ' όλα ε, το θέμα της Ισπανία. Δεν πρέπει να έχετε καμιά αμφιβολία όσον αφορά το 2012 και την ε, Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας. Καμία αφιβολία δεν πρέπει να έχετε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο, και η υποστήριξή της, η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι μόνο αποστολή των ε, διοικητών των ε, κρατικών εθνικών τραπεζών. Είμαι βέβαιος ότι στηρίζετε την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και δεν είστε ο κεντρικός τραπεζίτης. Οπότε το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και έπειτα, η Μπάνκη δεν διασώθη τον εγώ ήμουν υπουργό. Όχι. Υπήρχαν συγκεκριμένες συμμετοχικές ποσοστώσεις, δηλαδή μετοχές χωρίς οικονομικά δικαιώματα. Δεν έχει αυτό να κάνει με τις υπόλοιπες μετοχές. Έπειτα, ήμουν σύμβουλος ναι της BMN, αλλά επειδή ήμουν σύμβουλος, τα χρήματα αυτά ε, που είπατε για τη διάσωση της εν λόγω τράπεζας δόθηκαν πριν εγώ αναλάβω καθήκοντα. Και η αλήθεια είναι ότι ένα χρόνο που δούλεψα εκεί, πιστεύω πως συνέβαλα στην διάσωση και στην επιβίωση αυτού του θεσμού που θεωρώ πολύ σημαντικό. Και το θέμα της Μπάνκια. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι η Μπάνκια έπρεπε να εθνικοποιηθεί. Αλλά εκεί ποτέ εγώ δεν αναμίχθηκα, Ποτέ δεν είχε υπάρξει και τόση ανεξαρτησία όσον αφορά τη διαχείρισή τη. Δεν το λέω το λένε οι σημερινοί διαχειριστέ. Και η αναφορά που εσεί μου κάνατε αναφέρεται στην περίοδο πριν από την επανεθνικοποίηση. Και μάλιστα για μια κατάσταση πολύ περίπλοκη του ε, ισπανικού δημοσιονομικού συστήματο, μάλλον χρηματοπιστωτικού συστήματο, το οποίο είχε ενταχθεί πλήρω ευχαριστώ, Μάρκο eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω τι εξή ερωτήσει. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία τρίτου επίπεδου προ ε, την ρευστότητα του θεωρισμού. Υπάρχουν και άλλε παράμετροι όπω αυτή τη πλήρους απασχόληση σε όλε τι χώρε τη Ευρωζώνη. και ως εκ τούτου θα ήθελα να ρωτήσω πώ μπορεί μια κεντρική τράπεζα μόνη της να λύσει τις ανάγκες όσον αφορά τα ποσοστά της, του πληθωρισμού 19 οικονομιών που ε, έχουν πολύ διαφορετικές ε, πτυχές και εκφαλόγησης των, ε, των περιουσιακών στοιχείων τρίτου επίπεδου είναι αυτή όπου δεν διαπιστώνεται αξία στην αυτοκίνηση. Και άρα Θα πρέπει κατόπιν ε, εορτής ε, να γίνεται η αξιολόγηση και επαλήθευση. Εγώ ανέκαθεν θεωρούσα ότι η αξιολόγηση των ε, ενεργητικών των, των στοιχείων στην αγορά Πρέπει επίση να δούμε ποια είναι η δυνατότητα υπολογισμού των εσωτερικών με τα εξωτερικά μοντέλα. Πρόσφατα στη Βασιλεία επιτεύχθη μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία το output floor στόχος και εντολή της ΕΚΤ είναι σαφής, είναι αυτός του πληθωρισμού. Και αυτό περιλαμβάνεται, μπορεί να επηρεάσει θετικά το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών Μάλιστα, η νομισματική πολιτική λειτουργεί μέσω της αύξησης της συνολικής ζήτησης. Και αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών, αύξηση των πληθωρισμών και αύξηση τη δραστηριότητα. Και γι' αυτό και είπε και ο πρόεδρο Μπερντράγκη πω η νομισματική πολιτική ακολουθεί είναι, ε, μάλλον είναι αυτή που στηρίζει τη βελτίωση που είδαμε στην Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια. Δύο ερωτήσει να σα κάνω. Η πρώτη ερώτηση έχει φορά... Μιλήσατε για την ε, αρχή της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά δεν πιστεύετε ότι το δόγμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας ε, καθίσταται βασικό μελιάδος πρόβλημα της δημοκρατίας έναντι του Ευρωπαίου πολίτη. Όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, τις περιπτώσεις διαφθοράς στα Λετωνία, στην Κεντρική Τράπεζα και το καταστατικό της ε, Κεντρικής Τράπεζας δεν επιτρέπει να υποχρεωθεί κανείς να παραιτηθεί γιατί δεν μπορεί να κατηγορηθεί, να, να απαγγελθούν κατηγορίες. Άρα πιστεύετε ότι είναι φυσιολογικό ότι το δέχμα αυτό της ανεξαρτησίας ε, να κατοχυρώνεται έτσι ε, στην συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερη ερώτηση, θυμάμαι την εποχή της σύγκλησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για την ε, για το πολιτικό μείγμα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πολιτική. Ακούγοντα τι λέτε σήμερα, μου φαίνεται ότι θέλετε ακριβώς να δημορφώσετε αυτή τη μεικτή πολιτική στην Ευρωζώνη. Αυτό σκοπεύετε να κάνετε πολύ. Νομίζω πως η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών σύμφωνα με την οικονομική τεκμηρίωση ε, δείχνει ότι οι ανεξάρτητες ε, τράπεζες ε, δίνουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική δράση και την σταθεροποίηση του πληθωρισμού. Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, τα μοντέλα της νομισματικής πολιτικής βασίζονται στο monetary assessment και βεβαίως και όχι μόνο buffer αλλά και εξασφάλιση των καταθέσεων, εγγύηση των καταθέσεων. Θα μπορούσε να είναι ε, το bus stop της ε, ΟΝΕ και του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Εγώ που πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε μια ασφάλεια για την ανεργία. Θα ήταν πολύ καλύτερη λύση. Σε σχέση με το ε, ελεύθερο ενεργητικό που αναφέρατε, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα σφαιρικό θέμα είπε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι εκτός της βασιλείας, γιατί η τράπεζα, ο τραπεζικός τομέας είναι μια επιχείρηση παγκόσμια. Ε, ελεύθερο ενεργητικό κινδύνο. Τροποποιούμε τη δομή όλων των θεσμών που έχουν να κάνουν με το κίνδυνο. Είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα. Σε τρίτο επίπεδο, πιστεύω ότι για να σπάσει ο δεσμός ανάμεσα στις τράπεζες και την οικονομία δεν είναι τόσο θέμα του πόσο χρέος, δημόσιο χρέος έχουν οι τράπεζες στα για τους. Περισσότερο έχει να κάνει με τη μείωση του δημοσίου χρέους και του βάρους του δημοσίου χρέους σε σχέση με την οικονομία. Μακάρι το... 2012, αν οι τράπεζες είχαν ε, δημόσιο χρέας αντί να έχουν legacy assets, ίσως θα ήταν καλύτερα. Πιστεύω λοιπόν πως αυτό θα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, το του ESM. Για το Ταμείο Εξυγίασης. και για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει οι χώρες να αρχίσουν να διαπραγματεύονται. Είναι ένας βασικός πυλώνας της ε, μελλοντική Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που είχαμε με τον μηχανισμό εξυγίασης θα πρέπει να φτιάξουμε και να μπορέσουμε να έχουμε και ένα backstop, ε, αν θα είναι δηλαδή το, ο μηχανισμός σταθερότητας ή κάτι άλλο. Ε, πάντως θα πρέπει να αμοιβοποιηθεί το θέμα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Και έπειτα για προπολογισμό αντικυκλικό. Ε, θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τη συνένεση. Χρειαζόμαστε ένα προπολογισμό, χρειαζόμαστε ένα μέσο αντικυκλικό. Μπορεί να έχει διαφορετικέ μορφέ, μπορεί να είναι και η ε, δράση μέσω του κοινοτικού προπολογισμού ακόμα πρέπει να αρχίσουμε μια συζήτηση και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει μέσω μιας ασφάλειας για την, για την ανεργία. Όπως είπε η Ιταλική κυβέρνηση, η πρόταση της κυβέρνηση κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι δαπάνες για επενδύσεις. Αλλά πρώτα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποια είναι και αν είναι αναγκαίο ένα τέτοιο μέσο, ποιος θα το χειριστεί κατά τη γνώμη μου θα πρέπει αυτός να είναι η μελλοντική μορφή και σχηματισμός του ΙΣΕΜ και να υπάρξει και ευρωπαϊκό συντονισμό. Σας ευχαριστώ. Γκαμπριέλ Μάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διγκίντος για θέμα χρονοδιαγράμματος. Ε, είπατε ότι υπάρχει εγώ όχι. Δεν έχω καμία αφιβολία ε, για σας και, τη... και περνώ τώρα στην ερώτησή μου. Εσείς αναφερθήκατε στην ανάγκη να προχωρήσουμε στην Νομισματική Οικονομική Ένωση για να του δώσουμε το βάρος που χρειάζεται της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και μεγαλύτερης δυνατότητας να προβλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε τα ε, σοκ αυτά, Ε, πιστεύετε ότι θα αρκέσει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και έπειτα μιλήσατε ε, ότι για μείωση του ενεργητικού των μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων και στην Ισπανία αυτά μειώθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορούν αυτά να μειωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με τις τελευταίες προτάσεις της ΕΚΤ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μάτο. Σε σχέση με το θέμα του μέλλοντος της ε, ε, Νομισματικής Ένωσης, η Τραπεζική Ένωση ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι βασικό το να σχολιάσουμε πρώτα το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο γιατί είναι το τρίτο πόδι του τραπεζιού της Τραπεζικής Ένωσης. Δεν μπορεί να σταθεί ένα τραπέζι με δύο πόδια, θα χρειάζεται τουλάχιστον τρία. Και το τρίτο θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Και έπειτα, ε, ταμείο εξυπηρετούμενα δάνεια, για παράδειγμα, εγώ μίλησα για τη δημιουργία ε, ενεργητικού ή παθητικού, αυτή τη φορά δημιουργούνται από τις τράπεζες που έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης ε, ε, ζημιών. Δηλαδή, χωρίς να αγγίξουν τους καταθέτες και τους φορολογούμενους, αν μια τράπεζα έχει προβλήματα, να μπορεί να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βασική μου σκέψη πίσω από την μείωση του κινδύνου. Τώρα, σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα, ε, αυτό είναι ένα πολύ έδρο πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να αυξηθούν οι, οι ε, εγγύησεις και τα κεφάλαια των τραπεζών για να καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα 60 δις δημιουργία μιας κακής τράπεζας που θα μεταφερθούν όλα αυτά τα επιβαρημένα ενεργητικά, θα έχει αυτό το πλεονέκτημα που επιτρέπει στις τραπεζικές αρχές να επικεντρωθούν στα, στα ε, δραστηριότητε και να αφήσουν στην άκρη όλα τα αρνητικά και έχει να κάνει και με την ε, οδηγία για την ε, Είναι πολύ σημαντικό και είναι το βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Ταπεζικής Ένωσης. Αν υπάρχουν κίνδυνοι για συμμετρικά σοκ από πλευρά